Αγαπητοί συνάδελφοι, ξεκινάμε τη συνεδρίαση και το πρώτο σημείο της σημερινής ημερήσιας διάταξης είναι η ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και χαιρετίζω μεταξύ ημών τον κύριο Φιλίπ Μέιστατ, πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, ο οποίος θα συμμετάσχει στην σημερινή μας συζήτηση. Θα δώσω όμως καταρχήν για πέντε λεπτά τον λόγο στον εισηγητή. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι,